Συνταγματικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία και την Αφρική. συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα ταμεία. Εξ ονόματος του Συμβουλίου και πάλι ο Υπουργός, ο κ. Σμιτ. Παρακαλώ. Δουλεύει, μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά πόσο σοβαρή είναι η κρίση. Η κρίση την οποία εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Και είναι απολύτως ε, φυσιολογικό η κρίση, τα προβλήματα, οι δυσκολίες, αλλά και οι λύσεις να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχει λήξει η κρίση. Ούτε η κίνδυνη. Γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και η κατάσταση δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων επιδεινούται. Η Ευρώπη λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν παρέμειναν αδρανοί απέναντι σε αυτή την κατάσταση που θα τη χαρακτήριζα άκρος πολύπλοκη, γιατί εύκολες γρήγορες λύσεις σε αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχουν. Έγιναν ορισμένες προτάσεις, υλοποιούνται, ίσως υπερβολικά αργά, το παραδέχομαι, το λέω, όμως συμπληρωματικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα εξακολουθούν να είναι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη συνεδρίασή του της 23 Σεπτεμβρίου ανέλαβαν ορισμένες δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο ήδη από σήμερα για την Ευρώπη αποτελεί μείζωνα πρόκληση. Καταρχάς, θα πρέπει να στηρίξουμε τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ανάγκη από βοήθεια και που είναι πιο κοντά στη χώρα καταγωγής τους, ε, σε ε, καταβλισμούς. Με πάρα πολύ κακές, για να μην τις χαρακτηρίσω, είναι ότι καταστροφικές συνθήκες διαβίωσης. Συχνά δεν υπάρχει καμία σχολική εκπαίδευση για τα παιδιά, που είναι τα κύρια και τα πρώτα θύματα των συγκρούσεων αλλά και της κρίσης. Η ασφάλεια των τροφίμων σε αυτούς τους καταβλισμούς επίσης είναι επισφαλής ε, δύσκολη. Ξέρετε ποιες επιπτώσεις έχει. Έχει την φυγή των ανθρώπων αυτών προς την Ευρώπη, γιατί δεν έχουν πια καμιά άλλη επιλογή. Τώρα, είναι σημαντικό να τηρήσουμε τις δικές μας δεσμεύσεις, να τις εφαρμόσουμε, να τις υλοποιήσουμε. Η αύξηση ε, των συμμετοχών και των εισφορών των διαφόρων ανθρωπιστικών οργάνων ε, και οργανισμών, αλλά και ε, η ανθρωπιστική βοήθεια και έχουμε, είναι απαραίτητη και έχουμε και τα δύο αυτά καταπιστευματικά, καταπιστευματικά ταμεία για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι η αύξηση της υποστήριξης των διεθνών οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που στηρίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα την Πατεαρμοστή για τους πρόσφυγες και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι θα υποστηριχθούν με αυτά τα ποσά. Το μισό ε, θα προέρχεται από τον περιορισμό της Ένωσης και το άλλο μισό αυτής ε, τη ε, συμμετοχή θα είναι από διμερείς συμμετοχέ στι φορέ των κρατών μελών. Η πρώτη δέσμευση υλοποιήθηκε ήδη από τον Οκτώβριο. Τα κράτη-μέλη ανήγγυλαν ότι θα συνεισφέρουν με σημαντικά ποσά και μάλιστα θα ξεπεραστεί το 1 δισεκατομμύριο που προβλεπόταν και οι διμερείς συζητήσεις με τους δικαιούς οργανισμούς έχουν ήδη ξεκινήσει ώστε να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα προγράμματα αυτές οι δεσμεύσεις. Το ίδιο πράττει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα μας τα πει και η Επίτροπος. Σε ό,τι αφορά τα νέα ταμεία, τα δύο ε, καταπιστεύματα, Trust Fund, είναι σημαντικά εργαλεία που επιτρέπουν να συγκεντρώσουμε τα κονδύλια τα οποία προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πήγων από τον προπολογισμό τη Ένωση, από τα κράτη-μέλη αλλά και από τρίτε χώρε. Και από διάφορα κονδύλια του προπολογισμού, μεταξύ αυτών ανθρωπιστική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά τα ταμεία θα ανταποκριθούν στην κρίση της Συρίας και έχουν να κάνουν ε, με ε, την κατάσταση των ανθρωπιστικών οργανώσεων για την οποία σας μίλησα και την υποστήριξή της. Θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να τονίσουμε την ανάγκη σταθεροποίησης της κατάστασης. Η οποία είναι άκρος επισφαλής. Στην παρούσα φάση, οι συνεισφορές στο ταμείο αυτό, πρέπει να το ομολογήσουμε, δεν είναι ακόμη ικανοποιητική. Θα πρέπει να έχουμε αύξηση της συνεισφοράς μας, της συλλογικής συνεισφοράς μας, λόγω του ότι υπάρχει χρόνια υποχρηματοδότηση ε, των έργων που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον ΟΗΕ μόνο κατά 20%. 500 εκατομμύρια επιπλέον θα δώσουν τα κράτη-μέλη μέσω του προπολογισμού της Ένωσης. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει δεσμεύσει πάνω από 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη της κρίσης της Συρίας για την ανθρωπιστική δράση. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του ε, Συμβουλίου ε, υπενθυμίζει ότι όλα τα κρατη έχουν συλλογική ευθύνη. Τώρα, Αφρική. Ευθύνη δική μας είναι να δημιουργήσουμε βιώσιμες συνθήκες ώστε αυτοί που αναζητούν καλύτερη ζωή αλλού να έχουν ένα πιο αίσιο ε, ε, μέλλον και αισιόδοξο μέλλον στη δική τους χώρα για να ε, αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και την ενέργειά τους. Υπάρχουν διακινητές, εγκληματίες που παίρνουν χρήματα για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να πέρασουν στην Ευρώπη. Καλύτερα θα ήταν να επενδύσουμε αυτά τα χρήματα στην οικονομία της χώρας καταγωγής των ανθρώπων αυτών. Και για να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό δεν θα γίνει μια νυχτή και φυσικά και χρειάζεται μια νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη η οποία θα στηρίζεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων, στη δημιουργία εξωπρεπών θέσεων απασχόλησης στις αφρικανικές χώρες. Θα στηρίζεται σε επενδύσεις που θα κάνουμε ή θα στηρίζουμε σε αυτές τις χώρες, στην εκπαίδευση των νέων, που δεν επαρκεί πολλές φορές στην ανάπτυξη κλασικών κλάδων, οι οποίοι ενίοτε πλήττονται από έναν ανταγωνισμό και από την Ευρώπη στο επίπεδο της γεωργίας, της αλληλείας. Άρα έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε κάτι για το οποίο έχουμε αναλάβει και δέσμευση, δηλαδή να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη την ώρα που συζητούμε στη Μάλτα γίνεται η διάσκεψη κορυφής της Λαβαλέτα, όπου η Ένωση μαζί με τους Αφρικανικούς της εταίρους σκοπεύει να λάβει σημαντικές αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση. Και όπως μόλις προείπα, όταν λέμε μετανάστευση και όταν μιλάμε για μετανάστες, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα, τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Και το Ταμείο για τη Σταθερότητα ε, η καταπολέμηση επίσης της ε, λαθρομετανάστευσης, παράτυπης μετανάστευσης ε, είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Και βέβαια υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα. Δεν γίνονται βαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει καταπίεση, συγκεκριμένα φαινόμενα καταπίεσης. Αν δούμε πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι παράτυποι μετανάστες, πολλές φορές προέρχονται από χώρες όπου δεν υπάρχουν εγγύσει για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το αντίθετο μάλιστα ισχύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκής Ένωση στο Ταμείο της Αφρικής, θα υποδιαιρείται σε δύο τμήματα. Καταρχάς από το ΦΕΔ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κατά δεύτερον από τον προπολογισμό τη Ένωση. Εξού και ήταν δυνατό ήδη αυτής εξ αρχή να διευκρινιστεί αυτό, διότι θέλουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική και πρέπει να καλύπτουμε το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο διάστημα. Γιατί δεν είναι βραχυπρόθεσμο το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορεί να λυθεί παρά μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα διατεθούν κονδύλια της τάξης του 1,8 δις από τώρα μέχρι το 2020. Και πέραν τη σημαντικής αυτής συνεισφοράς μέσω του ΕΤΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη, που είναι διακυβερνητικό ταμείο, ακόμα ένα διακυβερνητικό ταμείο, σε αυτό το 1,8 δι προστίθεται η συμμετοχή από 20 τουλάχιστον ε, κράτη-μέλη που θα συνεισφέρουν σε εθνικό επίπεδο. Και η Νορβηγία έχει δηλώσει ότι θα συμμετέχει. Παράλληλα, έχουμε διμερά, προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών. Το καταπιστευματικό ταμείο είναι ένα στοιχείο της απάντησης, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον προγραμματισμό της συνήθους ε, βοήθειας που προσφέρουμε. Και νομίζω είναι ένας κοινός μας στόχος. Η διάσκεψη κορυφή τη Λαβαλέτα που είπε ότι λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή θα είναι η ευκαιρία να δοθεί αυτή η συμμετοχή ή επιπλέον. Βέβαια, σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω πιο ακριβή αριθμητικά στοιχεία, πιο οριστικά αριθμητικά στοιχεία για τις διμερεί συνεισφορέ στο κατεπήγον αυτό ταμείο, από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα εξαρτηθεί και από ε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Λαβαλέτα για αρκετά κράτη-μέλη. Να σας πω όμως ότι η δική μας χώρα, το Λουξεμβούργο, θα διαθέσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το καταπιστευματικό ταμείο. Έχουμε και 1,03% του ΑΕΠ που διαθέτουμε για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Υπενθυμίζω ότι όλοι έχουμε δεσμευθεί. Έχουμε δεσμευθεί εδώ και καιρό μάλιστα για 0,7% του ΑΕΠ. Και εντάξει, ίσως να μην περιμένουν όλο αυτό το 0,7%, δεν μπορούν να το πετύχουν. Η κατάσταση είναι τέτοια που ορισμένε χώρες μάλιστα μείωσαν την αναπτυξιακή τους βοήθεια. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική, αλλά ξέρετε ακόμα και στη δική μου χώρα φωνές ε, ζητούν να υπάρξει εξοικονόμηση σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ε, βλάπτει. Αλλά πρέπει, ξέρετε, να έχουμε υπόψη ότι ακόμη και στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και δημοσιονομικών περιορισμών η οικονομία, αυτή η εξοικονόμηση αυτή τελικά είναι κόστος. Διότι βλέπουμε ότι η μετανάστευση, η επανάπτυξη σήμερα είναι ουσιαστικά οι δύο του ίδιου νομίσματος. Και εάν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της πανάπτυξης, της εξαθλίωσης, του αποκλεισμού των νέων αναψώνες χώρες ε, με αποφασιστικότητα, κάποιοι θα το πληρώσουν με τη ζωή τους. Είπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι με φράχτες και, και σειρματοπλέγματα δεν θα αποφύγουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στο έδαφος ε, της Ανθρωπής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για μια επένδυση, ναι, σίγουρα στην αλληλεγγύη απέναντι στους γείτονες από την ε, Αφρική. Αλλά είναι και επένδυση στη δική μας την ασφάλεια. Και αυτό είναι η πρόκληση, αυτό διακυβεύεται εδώ. Και αυτό πρέπει σήμερα να πετύχουμε και να στείλουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη διάσκεψη της Λαβαλέτα. Ευχαριστώ. Ε, merci beaucoup, Monsieur Ministre. Now it's time for representative of European Commission. I'm ε, <coughs> sorry. Uh, Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Γεωργίευα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος μας έχει γίνει τόσο περίπλοκος και αλληλένδετος όπου παγκοσμίω ετησίως παράγονται 63 εκατομμύρια ευρώ και μέσα σε όλο αυτό το κόσμο ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζεται βοήθεια για να επιβιώσει αυξάνεται διαρκώς. 160 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται καθημερινή βοήθεια για να επιβιώσουν. Ήταν μια χώρα, θα ήταν η 11η μεγαλύτερη χώρα ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Τουρκία δηλαδή. Το μισό του πληθυσμού αυτής της χώρας είναι άστεγοι, εκτοπισμένοι λόγω ε, σειράξεων ή φυσικών καταστροφών και από αυτούς τους εκτοπισμένους το μεγαλύτερο μερίδιο ζει στη δική μας γειτονιά. Αφρική, Βόρειος Αφρική, Μέση Ανατολή. Και είναι σαφές ότι εμείς στην Ευρώπη δοκιμαζόμαστε όχι μόνο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ένα εκατομμύριο που τα κατάφερε να φτάσει στις ακτές μας, αλλά δοκιμαζόμαστε για να, να βοηθήσουμε 59 εκατομμύρια και αυτό το έργο είναι ηθικό σωστό, αλλά είναι και για το δικό μας συμφέρον. Αν θέλουμε να έχουμε πιο διαχειρίσιμη κατάσταση, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε όλο αυτό το κόσμο, πρέπει να αυξήσουμε την προσοχή μας και τη στήριξή μας για τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στην Τουρκία, αλλά και στις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Και γι' αυτό το λόγο εμείς στην Κομισιόν αποφασίσαμε ότι επιπλέον της, ε, της, της κανονικής μας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας θα χρησιμοποιούμε ένα νέο καταπίστευμα, ένα νέο μέσο που έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ε, κατά αποκοπήν ποσά που, κατα... που διαφορετικά θα ήταν πολύ μικρά και όχι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να λυθούν προβλήματα. Μας επιτρέπει να λάβουμε γρήγορα αποφάσεις ώστε να χρηματοδοτήσουμε δραστηριότητες και μας προσφέρει την ευελιξία ώστε να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Μας επιτρέπει δε να συγκεντρώσουμε περισσότερους δωρητές και έτσι να μειώσουμε το διοικητικό κόστος αλλά και να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας και τον ε, αντίκτυπο αυτού του μέσου. Πρόσφατα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε δύο τέτοια καταπιστεύματα. Το ένα είναι στην ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στην διάσκεψη κορυφής της Βαλέτα και θα ξεκινήσω με αυτό. Συζητήθηκε από την ύπατη εκπρόσωπα αντιπρόεδρο ε, Μογκερίνη και από τον Αντιπρόεδρο Μίμητσα ήδη στην ΑΦΕΤ και στην ΤΕΒΕ το Σεπτέμβριο στις 9 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Γιούνκερ ολοκλήρωσε την πρόεδρο αυτού του καταπιστεύματος με το στόχο να βοηθήσουμε ε, να αντιμετωπιστούν τα αίτια της αστάθειας και της ε, Άτακτη μετανάστευση, καθώς και να βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους πληθυσμούς στην Αφρική. Και με χαρά μπορώ να σας πω ότι από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ήδη είχε προχωρήσει η δουλειά με τρόπο ώστε να υιοθετήσουμε στην Κομισιόν τη σχετική απόφαση με ένα σχέδιο συντακτικής συμφωνίας ώστε να δημιουργηθεί ήδη αυτό το καταπίστευμα το οποίο εστιάζει την προσοχή στην παροχή οικονομικών ευκαιριών, τη στήριξη της αντοχής των ε, κοινοτήτων, την οικοδόμηση ε, ευκαιριών για ασφάλεια και ανάπτυξη καθώς και διαχείριση της μετανάστευσης στη Σαχέλ, στη κέρας της Αφρικής και τη Βόρεια Αφρική. Επίσης ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το τράστα μας επιστρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης αλλά και να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει άμεσες ανάγκες ε, προτεραιότητας. Είναι ευέλικτο, επιτρέπει τις άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες και επίσης είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο για περισσότερη ορατότητα της Ένωσης για το τι κάνει δηλαδή χρήματα δίνει. Ανάμεσα στις στοχευμένες δράσεις, πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε απασχόληση για τους νέους και για τις γυναίκες. Έχουμε, ε, οικοδομούμε δεσμούς ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ασφάλεια και στηρίζουμε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά τη μετανάστευση και τη διαχείριση των προσφύγων. Προσβλέπουμε στα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Βαλέτα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πλέον πόρους ε, σήμερα, όπως ακούσαμε και ε, από τον Υπουργό, έχουμε 1,8 δις στο καταπίστευμα αυτό, συν επιπλέον 70 εκατομμύρια που ήδη έχουν ε, υποσχεθεί τα κρατημέλη και ελπίζω πως θα δούμε και παραπάνω ε, τέτοιες ε, δεσμεύσεις στην διάσκεψη της Βαλέτα. Επίσης, να τονίσω ότι στο τράστ αυτό προτείνουμε την χορήγηση 200 εκατομμυρίων σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο για το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τινησία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω για ποιο λόγο αυτές οι χώρες αποτελούν ένα σημαντικό στόχο για τέτοιου είδους ε, ενίσχυση. Το δεύτερο καταπίστευμα που δημιουργήσαμε είναι το περιφερειακό καταπίστευμα για την ανταπόκριση στην κρίση της Συρίας. Δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 ώστε να ε, παρέχει πιο ε, ολοκληρωμένη βοήθεια σε περιφερειακή κλίμακα για τη Συρία καταρχήν ώστε να ε, καλυφθούν οι Σύριοι πρόσφυγες στις γειτονικέ χώρες. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τράστ επίση, ώστε να ε, βοηθήσουμε τους Σύριους που βρίσκονται στη Συρία αλλά και τους Σύριους που έχουν ήδη ε, ξεκινήσει την πορεία προς την Ευρώπη. και ορισμένες από τις χώρες από τις οποίες περνούν στη Δυτική στη, στη δυτική διαδρομή ε, και έχει, μάλιστα αυτό το καταπίστευμα ονομάζεται καταπίστευμα Μαντάτ με ε, σημαδιακό όνομα Μαντάτ σημαίνει ελπίδα Και αυτό επειδή πολλοί πρόσφυγες, πολλοί Σύριοι φεύγουν για την Ευρώπη επειδή έχουν χάσει την ελπίδα τους για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Ανάμεσα στους στόχους δε αυτού του καταπιστεύματος ε, είναι και η στήριξη της εκπαίδευσης ε, των παιδιών που είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Ήδη ο πόλεμος εκεί διαρκεί εδώ και πέντε χρόνια. Ήταν μια χώρα με πολύ καλές επιδόσεις στην παιδεία, 97 με 98% ε, ποσοστό αλφαβητισμού και όταν ε, ρωτούσε κανείς τα παιδιά τι ήθελαν να γίνουν όταν μεγαλώσουν, απαντούσαν γιατρός, μηχανικός, δάσκαλος. Τα δύο τρίτα τώρα από αυτά τα παιδιά είτε δεν πάνε καθόλου σχολείο, είτε πάνε πολύ κανόνιστα. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε ώστε να ε, εκπαιδευτούν όπως τους αξίζει, να βοηθήσουμε τις οικογένειές τους να μείνουν και να μην μετακινηθούν. ...που τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν και αυτά. Συν 32 δις, ε, εκατομμύρια. Και αυτά να τα δώσουν οι χώρες μέλη, αλλά ίσως και τρίτες και τρίτες χώρες. Ευχαριστώ τα κράτη-μέλη που ήδη συνεισέφεραν, αλλά και εκείνα που συνεισέφεραν όχι σε εμά αλλά στη UNICEF, ε, στο, στην Υπάτη Αρμαστία στο παγκόσμιο διατροφικό πρόγραμμα είναι το ΠΑΜ δηλαδή είναι για μας κρίσιμη αυτή η ώρα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο να δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη του καλού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπέ μου. Βλαγκοντάρια. Και τώρα οι εκπρόσωποι των πολιτικών αμάδων. Πρώτον, από το ΕΛΚ, Ράιμαρ Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, εγώ ακούω αυτά που επικαλείστε, αλλά έχω απογοητευτεί. Συμφωνώ στο εξής μαζί σας. Οποιο νομίζει ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα με σειρματοπλέγματα και τύχη, πλανάτε πλάνη ικτρά. Αλλά σήμερα δεν μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε ποιος, πότε και πόσο θα συνεισφέρει ε, σε αυτά τα καταπιστεύματα. Για να μην παρεξηγούμαστε, να εξηγούμαστε. Πριν από ένα μήνα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ε, επιγόντως ε, την κατάσταση για το 2015 και το 2016 9,2 δις με μαζικές μεταφορές πιστώσεων. Τα βρήκαμε τα λεφτά αυτά. Αλλά αν ακούσετε τι λέει ο Γκουτέρες που της είπα της αρμοστίας για τους πρόσφυγες 5.000 κάθε μέρα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, πάνω από 500.000. Δεν αρκούν αυτά τα μικρά σημεία. Ε, θέλουν να παραμείνουν σε καταβλισμούς κοντά στις χώρες τους. Και το παγκόσμιο επισητιστικό πρόγραμμα ακούμε τι γίνεται. Και τι κάνει η ύπατη αρμοστία. Και πόσα περισσότερα κονδύλια πήγανε. Μπορεί να είναι κάπως ε, μικρά τα ποσά, αλλά κινούνται. Αλλά δεν ε, έχουμε εξασφαλίσει την κατάσταση απέναντι στο χειμώνα που έρχεται. Και επίσης με το μηχανισμό κατανομής. Άρθρο Συγγνώμη, δύο λεπτά έχω, Πρόεδρε, και μην με πιέζετε. No, two minutes. Uh, uh, two minutes. Two minutes ε, δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Συν δεκαδεύτερα που με διακόψατε. Λοιπόν, άρθρο 78, εδάφιο 3, όχι, δεν θα πρέπει να είχε χρησιμοποιηθεί αυτό το άρθρο, αλλά θα έπρεπε να είχαμε ε, ε, καταφύγει στο άρθρο 97.3 για κοινή ρύθμιση για την προσωρινή προστασία όταν έχουμε μαζική είσοδο. Αυτό όμως δεν το τολμήσαμε και πολλά κράτη εκεί είναι συνυπεύθυνα. Έχω λοιπόν την εξή παράκληση. Πραγματικά σας συγκετεύω να ε, λειτουργήσει αυτή τη λύση του καταπιστεύματος, αλλιώς θα πρέπει να την αφισβητήσουμε. Και κυρία Επίτροπη, να δίνεται έκθεση σε κάθε ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ποιος, πόσα και πότε, αλλιώς θα χάσουμε ακόμα και την ελάχιστη αξιοπιστία που μας έχει απομείνει. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ε, ε, Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. κάποιο λάθος έγινε, μια παρεξήγηση, γιατί εδώ στα χαρτιά μου λέει ότι έχετε 1,5 λεπτό. Εντάξει, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σας και με χαρά να σας δώσω και δυόμιση λεπτά. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχει η κυρία Γουαριαθάμπαλ Ρούμπια. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω την κατάσταση των προσφύγων που ζούμε και την πρόκληση που συνιστά αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, νομική, κοινωνική, ανθρωπιστική και δημοσιονομική πρόκληση. Σε αυτό το τελευταίο θα σταθώ. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε το θεματολόγιο για το προσφυγικό, είχε συμπεριλάβει περίπου 17 δισεκατομμύρια και μεταξύ αυτών είναι τα 2-300 για το καταπίστευμα για την Αφρική και την Σύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά κάνει αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την κρίση. Αλλά οι ανάγκε και οι δεσμεύσει δεν σταματούν εκεί. Αυτόν ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τι γίνεται όμω με εκείνον που αντιστοιχεί στους κρατικούς προπολογισμού. Και το άτυπο συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, το θύμισε ο, επι, ο Υπουργός ε, Σμιτ, ε, είδε τα κράτη-μέλη να δεσμεύονται για το παγκόσμιο επισητιστικό πρόγραμμα για την υπατιαρμοστία πάνω από ένα δις, πέρα από την ευρωπαϊκή συνεισφορά. Και παρόλα αυτά και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν κάποιες χώρες, μας λείπουν πάνω από δύο δις. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά. Βέβαια όλα τα νέα δεν είναι κακά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 9,4 δις με διάφορες προσαρμογές αλλά και εκτάκτους πόρους και έσοδα από πρόστιμα και δασμούς. Ωραία, τα είπαμε αυτά στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν αφισβητεί ούτε τα, τα ποσά, ούτε την νομιμότητα, ε, αλλά θα ήταν επίσης αξιέπαινο πολιτικό ε, μήνυμα 28 να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα αυτών των κονδυλίων για να χρηματοδοτήσουν εκείνα που τους αναλογούν στο καταπίστευμα. Θα πρέπει τα έργα μας να συμφωνούν με τα λόγια και τις δεσμεύσεις μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία που δεν επιτρέπεται να ε, αποτύχουμε. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έτσι κατέληγαν οι τρεις ε, πρόεδροι στους 28 στην επιστολή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ε, ο κύριος Κόλμελ. Και θα προσέχω περισσότερο το χρόνο να το τηρείτε. Να, μισή λεπτό. Όλοι καταλάβαμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της σημερινής κρίσης θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και μεταξύ αυτών ανήκει και η συμφωνία στην αίτηση αυτή, γιατί και η Συρία και η σύνολη Αφρικανική πυρός χρειάζονται τώρα ακριβώς τη βοήθειά μας. Γι' αυτό 2,3 δις είναι ένα καλό ποσό. Το ξέρω ότι δεν επαρκεί, αλλά τι να κάνουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο απαραίτητο και αναγκαίο από δημοσιονομική σκοπιά, αλλά και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο τα χρήματα αυτά να πιάνουν τόπο. Θα πρέπει λοιπόν να τα δαπανούμε όσο γίνεται πιο κοντά στις αιστείες ανάφλεξης και κρίσης, γιατί εκεί πιάνουν τόπο ακριβώς, γιατί εκεί με λιγότερα χρήματα ή με τα ίδια χρήματα μπορούμε να πετυχάνουμε περισσότερα. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να φεύγει στην προσφυγιά και να κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι να σωθεί. Θα πρέπει να τους βοηθάμε όσο γίνεται πιο κοντά στην πατρίδα τους. Το σημερινό μας θέμα είναι ο προπολογισμό. Αλλά αυτό που πάντα εμείς... Ε, στιγματίζουμε είναι μόνο για λεφτά συζητάμε και για προϋπολογισμό. Δεν συζητάμε γενικότερα για τη συνολική εικόνα και θεώρηση που να είναι και στο ύψος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε κάποια στιγμή να δούμε συνολικά, σφαιρικά τα προβλήματα αυτά και να φέρουμε ουσιαστική λύση. Η κρίση αυτή δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με λεφτά. Χρειάζονται τα χρήματα αλλά δεν αρκούν. Είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι αρκετή. Θα πρέπει να ο νόμος και ε, στην Ένωση και να χρησιμοποιούνται όλα αυτά σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Σας άκουσα με προσοχή και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι ήθελα κι άλλα η σοβαρότητα της κατάστασης ε, την χάνει κάποιας ε, υποτίμησης εδώ. Τρία παραπάνω εκατομμύρια πρόσφυγες θα έρθουν τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε. Και αυτά που αναμένετε ως αποτελέσματα από τα μέτρα που θα λάβετε επίσης είναι λίγο απογοητευτικά. Ένα δις για τη Συρία. Αν τα κράτη-μέλη βάλουν τα 500 εκατομμύρια που έχουν υποσχεθεί είναι τα 500 της Κομισιόν ενώ υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και ένα ακόμα παραπάνω μέσα στη Συρία 160.000 πρόσφυγες θα έχουμε στην Ευρώπη και θα δαπανίσουμε ένα δις σύνολο. Από αυτό το δις ανα, μήπως αναμένεται υπερβολικά πολλά. Τι έχει ήδη εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο η διμερή συνεργασία. Ένα δις για το Συριακό Ταμείο το Αφρικανικό αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι αφελές να πιστεύετε ότι κάτι πρόκειται να γίνει με αυτά η Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν μια σφαιρική στρατηγική και μετά να συνδυάσουν όλα τα εργαλεία που διαθέτουν, να δουν τι μπορούν να κινητοποιήσουν για να υπάρχουν, υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι μέχρι τώρα. Σε ποιον λοιπόν θα δοθούν αυτά τα λεφτά για την Τουρκία, α πούμε, στον Ερντογάν ή σε οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Συνεργασία. Ναι, αλλά όχι δουλεία. Η κυρία Ριάδα. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να προσπιστούμε την αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για να τονίσουμε, να στηρίξουμε όλες αυτές τις ε, προσπάθειες και μάλιστα σε διαφανές πλαίσιο. Χαιρόμαστε για τη διαφάνεια, αλλά τα ταμεία αυτά δεν έχουν πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα που πρέπει σε χώρες όπως τη Συρία, την Τουρκία ή ορισμένες περιοχές της Αφρικής. Καμιά φορά επενδύουμε παραπάνω μου φαίνεται για κτίρια και έπιπλα παρά στα καταπιστεύματα αυτά για την Αφρική ιδίως. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να διασφαλίσει ότι ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση θα έρθει να απαντήσει σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για αυτά τα καταπιστεύματα καθώς και για θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Πρέπει να διατεθεί πλήρης πληροφόρηση για το ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για αυτά τα σχέδια και προγράμματα, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι θα σέβονται απολύτως τους κανόνες της Ένωσης, να βελτιωθούν τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να είναι πιο ευέλικτα, ώστε να είναι σαφές ότι θα υπάρχει διαδικασία διαφανής και δημοκρατή. Η κυρία Χάουταλα για δύο ολόκληρα λεπτά. Πρόεδρε, θυμάμαι πολύ καλά όταν η Επίτροπος Γεωργίευα έκανε την τελευταία της επίσκεψη στην Επιτροπή Ανάπτυξης πριν να γίνει αντιπρόεδρος υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι κυρία Γεωργίευα μου είχατε πει ότι αν δεν λυθούν οι ρίζες, οι λόγοι της ανθρωπιστικής κρίσης, κανείς δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις τους όπως θα συνεχίζονται. Φυσικά είχατε δίκιο και είδαμε ήδη τι συμβαίνει. Επίσης πρέπει να πω ότι χαίρομαι που είναι παρούσα και η Λουξεμβουργική Προεδρία εδώ, διότι το Λουξεμβούργο είναι μικρός αλλά πολύ συνεπής δωρητής. Να μην τρέπεστε για τις μειώσεις που κάνουν άλλες χώρες μέλη στις εισφορές τους για τα ανθρωπιστικά. Ντρέπομαι ιδιαίτερα που η Φιλανδία μειώνει το μερίδιό της κατά 42% σχέτη καταστροφή. Ο δε πρόεδρος Γιονκέρ είπε ότι δεν είναι φυσικό να κόβουν χώρες μέλη ...τον αναπτυξιακό του, στον προϋπασμό του για την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχω όμως τώρα μερικά ερωτήματα και απορίες. Όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κατεπίγουσες καταστάσεις, πώς θα σεβαστούμε την αρχή της αποτελεσματικότητας της ανάληψης των καθηκόντων από την ίδια τη χώρα που επωφελείται γιατί ξέρετε ότι ποια είναι τα προβλήματα. Τα χρήματα αυτά δεν είναι καινούρια βέβαια και πρέπει να καταλάβουμε ότι θα χρειαστούν να περικοπούν ορισμένες δραστηριότητες για να δοθούν τα χρήματα σε αυτές. Πώς θα συμπληρωθούν λοιπόν αυτά τα καταπισουτεύματα, πώς θα συνδυαστούν με τις υπόλοιπες σας κατευχαριστώ. Κοράω. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τόσο ο πρόεδρο τη Επιτροπή Γιούνκερ, όσο και είπα ότι εκπρόσωπο Μογκερίνη, αλλά και η Επίτροπο Γεωργίευα, επανελειμμένω υπογράμμισαν τη, την σημασία τη αντιμετώπιση τη ε, μετανάστευση και τα βαθύτερα αίτια τη, ε, θυμίζοντα επίση τη δέσμευση των κρατών μελών. Η πραγματικότητα όμω, κατά την εντύπωσή μου, είναι, η εντύπωσή μου είναι, ε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Διαντρέ, ότι η Ευρώπη χωρί καμιά αξιοπρέπεια κάνει πω νοιάζεται και μετά στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Στην πραγματικότητα δεν γίνονται σεβαστές οι δεσμεύσεις, είναι λόγια τα οποία δεν ακολουθούν ε, πράξεις. Τώρα, μιλώντας για αυτό το καταπίστευμα, γνωρίζουμε ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία μετακινούνται από την αναπτυξιακή βοήθεια. Οπότε, κινδυνεύουμε να έχουμε μία... ε, ε ένα αποτέλεσμα όπως η μεθαδόνη για τους ναρκωμανείς. Δηλαδή ε, δεν λύνουμε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε αυτά που οδηγούν στην μεγάλη μετανάστευση. Πρέπει να παρέμβουμε με σοβαρά προγράμματα βοηθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παιδεία και την υγεία. Ο κύριος Μπέι, επόμενος ομιλητής, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μάθαμε σήμερα ότι ο Συριακός Σταθμός κατάφερε να συντρίψει την αντίσταση που του αντιστεκόταν γύρω από το Χαλέπι, τη μαρτυρική αυτή πόλη. Χαιρετίζω την νίκη αυτή κατά του Ισλαμικού κράτους και εύχομαι να επρόκειται για την αρχή του τέλους εδώ, για αυτή την τρομοκρατική οργάνωση. Από την αρχή της σύραξης στη Συρία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έδειξαν έλλειψη ρεαλισμού ρίχνοντας λάδι στη φωτιά, κλείνοντας τις πρεσβείες τους και υποστηρίζοντας την αντιπολίτευση που ε, δεν είχε τίποτα το δημοκρατικό. Η επανάληψη των δημοκλωματικών σχέσεων με τη Συρία θα ήταν μία προϋπόθεση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εδώ πρόκειται επιτέλους για κάποια λογική από την Ένωση. Εξάλλου αυτό θα ήταν το λογικό όπως έκαναν ορισμένες άλλες φορές να μην έχουμε διακόψει ποτέ τις διπλωματικές μας σχέσεις με τη Συρία. Όσο για τη βοήθεια προς το Συριακό λαό λυπάμαι γιατί στοιχηματίσατε σε οργανώσεις όπως τους γιατρούς χωρίς σύνορα οι οποίοι παρεμβαίνουν μόνο στις περιοχές όπου βρίσκονται οι αντάρτες. Ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ που πήγαιναν και αλλού δεν έχουν σήμερα χρηματοδότηση. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως το SOS Χριστιανοί της Ανατολής αποδείχτηκαν πολύ πιο θαραλέε και αποτελεσματικές όχι μόνο στη Συρία αλλά και στο Λίβανο και αλλού. Κάνουν καταπληκτική δουλειά χάρη στο διάλογο που δημιούργησαν με τις τοπικές αρχές. Εμπνευστείτε λοιπόν από αυτό το ρεαλισμό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βαλτσόχνερ γεγραμμένος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Για να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε την κρίση των προσφύγων θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι τα αίτια για να καταλάβουμε. Γι' αυτό κατά πρώτο λόγο χρειάζεται διεθνή συνεργασία με τις χώρες ε, της Αραβικής Άνοιξης. Η σημερινή απόφαση ίδρυσης των καταπιστευμάτων αυτών είναι πολύ σημαντική και θετική και έτσι θα καταφέρουμε να βοηθούμε τους πρόσφυγες κοντά στην πατρίδα τους και να παραμένουν εκεί. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να φροντίσουμε τα σύνορα του Σέγγεν στην Ελλάδα συγκεκριμένα να προστατεύονται και να φυλάσσονται. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, το μόνο που μπορούμε ε, να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε μεθόδους τύπου Ουγγαρίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την κρίση αυτή την προσφυγική και να προστατεύσουμε την ταυτότητα και την ακαιρεότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνονται εδώ οι ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και ακολουθούν μεμονωμένοι βουλευτές. Πρώτος ο κύριος Φερνάντης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη θα λάβουν τώρα στα τέλη του έτους 9 δις 400 ε, εκατομμύρια από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έσοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί ε, και έκτακτα έσοδα δηλαδή. Ε, δύο δις από αυτά είναι έσοδα από πρόστιμα και από τελωνιακά τέλη είναι ένα ποσό που τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν στα καταπιστεύματα για τη Συρία και την Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς καμία επιπλέον οικονομική βοήθεια, χωρίς να ψάξουν, να προσπαθήσουν και να πιέσουν τους προϋπολογισμούς τους, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δύο δις 300 εκατομμύρια ευρώ για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στις δύο αυτές υποθέσεις. Αυτή η υποχρέωση των απέναντι στους πρόσφυγες, ε, αυτή η προσφυγική κρίση όπου τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν στην ε, ρίζα τους και όπου πρέπει όλοι να συμμετέχουν για την επίλυσή τους, αυτά τα δύο καταπιστεύονται θα δώσουν ελπίδα, θα δώσουν εγγύησεις για ένα καλύτερο μέλλον, θα συμβάλλουν για την παιδεία, για την ε, εκπαίδευση των ανθρώπων στη χώρα τους, να προλάβουν και όχι να θεραπεύσουν. Πάντα είναι αυτό καλύτερο και ελπίζω ότι αυτά τα ποσά, τα επιπλέον, που ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιστρέψει στου εθνικού προπολογισμού, ελπίζω να χρησιμοποιηθούν για να, να βοηθήσουν μάλλον στη λύση αυτού του προβλήματο. Ευχαριστώ. Κύριε Φερνάντε, υπάρχει μια αλλάζια κάρτα από τον κύριο Κόμπορν. Τη δέχεστε? Μάλιστα. Κύριε Κόμπον, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω μια ερώτηση τον κύριο εδώ για να δω αν συμφωνεί μαζί μου. Μήπω δεν ήταν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή η Μεγάλη Βρετανία έχει βάλει περισσότερα χρήματα για του καταβλισμού στα Συριαοτουρκικά σύνορα από οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα ήταν καλύτερα αν αυτέ οι χώρε έδιναν τα χρήματα οι ίδιε ή έφτιαχναν του δικού του καταβλισμού στη Συρία παρά να παίρνει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα σπαταλήσει ε, με τον συνήθι τρόπο. Νομίζω πως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν ελέγξει σωστά τους λογαριασμούς εδώ και 20 χρόνια. Ας τα κάνουν λοιπόν μόνη της η κάθε εθνική κυβέρνηση και να μην απ' έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα αυτά. Κύριε Φερνάντες, παρακαλώ να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι τα κάτι μέλη θα λάβουν επιπλέον χρήματα. Άρα λοιπόν είναι στη δική του διακριτική ευκαιρία και στη βούλησή του να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για αυτό το στόχο. Εγώ αυτό που πρότεινα είναι κανένα φορολογούμενο από καμιά χώρα με αυτά τα χρήματα που είναι επιπλέον έσοδα από, από πρόστιμο και από τελωνιακά τέλη δεν θα χρειαστεί να συμβάλλει ώστε να ε, ε, ε, με παραπάνω χρήματα. Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά, να τα διαχειριστούμε σωστά, οι στόχοι να επιτευχθούν και να χρησιμοποιηθούν με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είναι προφανές ότι πάντοτε αυτό δεν το καταφέρνει οποιοδήποτε κράτος και οποιοδήποτε ε, οργανισμός μπορεί να μην τα καταφέρει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάιερ. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Σμιτ, κύριε Αντιπρόεδρε Γεωργιέβα, ας φανταστούμε μια στιγμή έναν ασθενή στον τιβάνι ενός ψυχιάτρου που λέει περίπου αυτά. Γιατρέ, είμαι πρωθυπουργό κράτου μέλου Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είμαι στι Βρυξέλλε με του συναδέλφου μου εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άνδρε και γυναίκε, αποφασίζω ε, πράγματα που ζητώ ως ε, ε, Πρωθυπουργό να δοθούν χρήματα στα ταμεία αυτά για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Μετά γυρνάω στο γραφείο μου, ε, στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και λέω καλά αυτά είναι δηλώσεις προθέσεων και δεν είναι δεσμευτικά ε, και αυτή την απέτηση την αγνοώ. Τι θα έκανε ο ψυχίατρος, θα μου γράφε φάρμακα, θεραπεία σίγουρα. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ανέκδοτο, αλλά είναι πραγματικότητα στην Ευρώπη. Έτσι συνεδριάζει το Συμβούλιο. Σωστά συνιστά να γίνουν καταπιστεύματα για να καταπιστευθεί η κρίση, αλλά τα κράτη-μέλη δεν δρούν επαρκώς, δίνουν πενταροδεκάρες. Και αυτή είναι μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη ε, δεν δρούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ε, τον προπολογισμό το διορθωτικό 8-2015 έχει βρει 9 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν χρήματα λοιπόν, είναι σχεδόν 100 φορές περισσότερα από τα 82 εκατομμύρια ε, που θέλει να δώσει το Συμβούλιο το 16. Και λέει, ε, γιατί υπάρχει δυνατότητα έτσι να αντιδράσουμε σε απρόπτα. Παρακαλώ το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που έχει η Πρόεδρος Διακόπτη τον ομιλητή για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση, αλλιώς θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οζόκα, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν ε, για τα καταπιστεύματα έχει στόχο να διαχειριστεί καλύτερα και τις ε, μεταναστευτικές ροές. Ένωση λοιπόν ήδη έχει δεσμευτεί για ψηλά ποσά αλλά περιμένει από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν και εκείνα. Μέχρι τώρα πολύ λίγα το έπραξαν. Ερωτώ λοιπόν. Τι θα κάνει η Κομισιόν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και έπειτα. Μερικές χώρες μέλη εξών και η Πολωνία θέλουν να δεσμευτούν και για άλλα προγράμματα όπως το Παγκόσμιο Διατροφικό Πρόγραμμα. Επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα συνδυαστούν αυτά τα καταπιστεύματα με τα υπάρχοντα εκείνα προγράμματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το καταπίστευμα για τη Συρία στοχεύει στα παιδιά και του νέους και την παιδεία, την επιβίωση και την ε, διατροφική ασφάλεια. Όμως για την Αφρική πρέπει να καταπολεμηθούν οι βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης, δηλαδή να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία της χαρτούμα σε συνεργασία με τις χώρες ε, όπως το Σουδάν που εξακολουθεί να ε, βομβαρδίζει τον πληθυσμό του, 3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Ερυθρέα επίσης όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά. Αυτές οι χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το 1,8 ε, δις θα πρέπει να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Οι Αφρικανοί αρχίζουν να λένε ότι δεν θέλουν να κάνουν τους αστυνομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινησμός, ε, όνειρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφει τα νότα στο καθήκον της για την ανθρωπότητα. Πολλοί εκτοπισμένοι, πολλά εκατομμύρια Αφρικανοί είναι εκτοπισμένοι εντός της Αφρικής. Ευχαριστούμε. Κυρία Βαλέρο. Κυρία Βαλέρο, 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Οποιαδήποτε ζωή χάνεται στον δρόμο για την Ευρώπη είναι πολύ υπερβολική. Είτε ξεφεύγει κανείς από τη Συρία και τον πόλεμο είτε από τη φτώχεια στην Αφρική. Όπως είχε πει και ο Σμιτ, δεν πρόκειται να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ούτε οι πρόσφυγες, ούτε οι μετανάστες. Που ζη... Για όσους ζητούν δηλαδή να επιστραφούν, αυτοί θα ξανάρθουν. Αν δεν λυθούν οι ουσιώδεις λόγοι, οι ρίζες του προβλήματος. Και εδώ πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσαμε Διαβάζω την απόφαση του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου και βλέπω ότι δίνεται πολύ σημασία στη μετανάστευση και στο σταμάτημα των ανθρώπων στα σύνορα. Τίποτε πιο μακροπρόθεσμο όμως ώστε να υπάρξουν να υπάρξει περισσότερη ανάπτυξη ας πούμε στις χώρες προέλευσης. Έτσι βέβαια δεν δίνουμε χρήματα ούτε και σε προγράμματα τέτοια μακρόπνοα. Επίσης, στον προϋπολογισμό είπαν πολλοί ότι οι χώρες μειώνουν την εισφορά τους για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών γιατί αυτή θεωρείται και αυτή ένα είδος αναπτυξιακής βοήθειας idea of dealing with the problems of mass migration at source or as close. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την μαζική μετανάστευση ε, στην ε, πηγή της. Αυτό είναι πρόσδεκτο. Θέλουμε να δοθούν παγκόσμιες λύσεις στις χώρες προέλευσης ή στα γειτονικά κράτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά ενώ το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει άλλη μια κρίση για να ζητήσει περισσότερα χρήματα από τους ξεζουμισμένους Βρετανούς φορολογούμενους, εμείς λέμε όχι. Ε, δεν έχει νόημα το να υπάρχουν αρκετά χρήματα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να αρχίσουμε να σπαταλούμε τα χρήματα, μάλλον να πάψουμε να σταματούμε αυτά τα χρήματα σε μη ουσιαστικά προγράμματα ε, και τα τοποθετήσουμε σε προγράμματα πραγματικά με νόημα, μπορεί το κοινό να αρχίσει να πιστεύει πάλι σε εμά. Ε, χαλάμε δισεκατομμύρια σε διάφορα εκπαιδευτικό υλικό ε, χωρίς κανένα λόγο. Αντί να προωθούμε τις αξίες μας μέσα από την προπαγάνδα, καλά θα ήταν να δίνει το παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματώντας να πανά αυτά τα χρήματα άσκοπα και κατευθύνοντάς τις σε ουσιαστικά ε, θέματα όπως την επίλυση της προσφυγικής κρίσης. Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, κυρία Πίτροπε, τη Δευτέρα συναντήθηκαν εκτάκτως Υπουργοί Εσωτερικών και πάλι με αποτέλεσμα ε, να ευαισθητοποιηθεί, λέει, η κοινή γνώμη και τα κράτη-μέλη. Αυτά δεν ε, επαρκούν. Είναι τεράστια η κρίση ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δεν επαρκούν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζουν τίποτα με βιώσιμο τρόπο. Δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Frontex δεν έχει αρκετά ε, μέσα στη διάθεσή της και τελείως ε, τεράστια εντολή. 160.000 επανεκαταστάσεις και μετεκαταστάσεις ε, δεν βοηθούν. Δεν αρκούν όλα αυτά. Και τα σημερινά κονδύλια που τάζουμε μπορεί να τα καλωσορίζω και τα καταπιστεύματα, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πότε, πόσα και ποιος θα τα δώσει αυτά τα πράγματα είναι αφόρητα. Πολλοί ε, έχουμε καθυστερήσει. Εδώ και ένα χρόνο μας λένε το παγκόσμιο επισητιστικό πρόγραμμα, η πατιαρμοστία, το ταμείο είναι μείον και εμείς κοφεύουμε. Τι θα γίνει, πώς θα λύθει αυτή η κατάσταση. Πάνω από 400.000 πρόσφυγες ε, που έχουν διακινηθεί. Είναι αφόρητη η κατάσταση και η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ο κύριος Επιτίδιος, παρακαλώ. Ένα λεπτό. στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως ε, του προβλήματος που προέκυψε λόγω της κρίσεως στη συρία αλλά και των αιτίων ε, μεταναστεύσεως και μετακινήσεως στην αφρική τα κράτη της ευρωπαϊκής ενώσεως θα υποχρεωθούν να καταβάλουν περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. πλανόμαστε όμως πλάνη νυχτρά, εάν νομίζουμε ότι με τα χρήματα αυτά θα επιλύσουμε το πρόβλημα οι μετανάστε και οι πρόσφυγε θα εξακολουθήσουν να έρχονται κατά κύματα στην ευρώπη η ανάγκη χρηματοδοτήσεώ όσο θα εξακολουθήσει να υπάρχει και οι λαοί τη ευρώπη και ιδιαίτερα ο πολύπαθο ελληνικό λαό θα εξακολουθήσουν να υποφέρουν από τα εξοντοτικά μέτρα λιτότητα που επιβάλλονται για να χρηματοδοτούνται οι παράνομοι μετανάστε. για να αντιμετωπίσουμε μερικώς το πρόβλημα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσβάλλουμε τα αίτια τα οποία το προκάλεσαν θα πρέπει να σταματήσουν καταρχά οι πόλεμοι που διεξάγονται στι χώρε αυτέ. επίση τα χρήματα θα πρέπει να δίδονται στι χώρε προελεύσεω των μεταναστών ούτω ώστε να αναπτυχθούν οικονομικά αυτέ και να μην επιτρέπουν οι κυβερνήσει τη μετανάστευση προ την ευρώπη. τα κέντρα ελέγχου και ταυτοποίηση τα hot spots θα πρέπει να γίνονται στι χώρε προελεύσεω και όχι στι χώρε εισόδου. και τέλο θα πρέπει να υποχρεωθεί η τουρκία να πάψει να στέλνει κατά χιλιάδε πρόσφυγε προ την ελλάδα και την ευρώπη. The uh, Επόμενος ο κύριος Στίερ. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ήθελε μια σφαιρική λύση του προβλήματος των μεταναστών και γι' αυτό δεχόμαστε τα δύο νέα καταπιστεύματα. αν θέλουμε επικοδομητικές συζητήσεις στη Βαλέτα καθώς και τις επιστροφές στις χώρες προέλευσης των μεταναστών που δεν θα έχουν γίνει δεκτοί. Τότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιδείξουν τη θέλησή τους να συμμετρησότερο ιδιαίτερα γιατί ακούστηκε ο αριθμός του 1,8 δισεκατομμυρίου που θα πρέπει να περικοπούν από αλλού πρέπει να τονίσουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας και αναμένουμε κυρία Επίτροπε να μας δώσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των κοντιλίων για να μην γίνουν καταστούν, καταντήσουν άλοθη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε και το χρόνο σας η κυρία Τεμά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκφραση αυτή του κυρίου Γιούνκερ θα μας ακολουθεί πολύ καιρό, ότι είμαστε αναγκασμένοι δηλαδή να φταρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία αυτών των δύο καταπίσου τεφουμάτων. Όμως υπάρχουν και δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι οι χρηματικές υποσχέσεις των κρατών μελών που δεν τηρήθηκαν και δεύτερον ότι το ανώτα, τα τα όρια των σχετικών θέσεων του προπολογισμού είναι πολύ χαμηλά και δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Άρα χρειάζεται να βρει, βρει η Κομισιόν πόρους εκτός προϋπολογισμού και άρα χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Είναι λοιπόν ο προϋπολογισμός πνίγεται. Η κρίση θα συνεχιστεί και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και άλλες κρίσεις. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δημοσιονομική πραγματικότητα ως έχει. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, το έχουμε πει και άλλη φορά στην αίθουσα αυτή. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλημμυρίσει από τους χιλιάδες δύστιχους πρόσφυγες της Συρίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει τελικά. Δίνει ψίχουλα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στη φτωχοποιημένη από τα μνημόνια Ελλάδα. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θοπεύει την Τουρκία αντί να την απειλήσει με λήψη μέτρων αν δεν σταματήσει τα δουλεμπορικά κυκλώματα που δρούν ανεξέλεγκτα μεταφέροντας χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες στο αιγαίο. πρέπει λοιπόν πρώτον τα hot spots να δημιουργηθούν στην τουρκία και σε άλλες τρίτες χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης. δεύτερον να καταργηθεί το δουβλίνο τρία και να εφαρμοστεί η ρήτρα κατανομής προσφύγων και παράνομων μεταναστών σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης ανάλογα με το αεπ τον πληθυσμό και την έκταση κάθε χώρας τρίτον να δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια στις χώρες της αφρικής για να σταματήσει η από εκεί παράνομη μετανάστευση. τέλος να ενταθούν οι προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της συριακής κρίσης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Α, δουλεύει, δουλεύει. Α, ευχαριστώ πολύ. 1,3 εκατομμύρια ε, μετανάστες και πρόσφυγες ήρθαν φέτος, αναμένονται τρεις του χρόνου. Ε, και τι κάνει η Ένωση, ένα καταπίστευμα, ένα-δυο ε, δισεκατομμύρια για να λύσει μαζί και το αφρικανικό λέει πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε γιατί υποστήριξε τις καθεστωτικές αλλαγές στη Λιβύη και αλλού και δημιουργήθηκε επίσης γιατί δίνονται άδικοι φόροι και δεσμοί σε προϊόντα από την Αφρική. Η Ένωση δεν είναι φίλος της Αφρικής ούτε των Αφρικανικών λαών. Δεν είναι φίλος των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει η Ήπειρος αυτή για ανάπτυξη. Η Ευρώπη εφαρμόζει απικιακές ακόμη πολιτικές. Η αδυναμία της Αφρικής να ταΐσει τους λαούς της μόνη της, να τους θρέψει, δεν χρησιμοποιούνται γιατί η μόνη προσπάθεια που γίνεται είναι πώς θα εξαχθεί καφές στη Γερμανία. Είπαμε πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να τους δίνουμε ψάρια αλλά να τους διδάξουμε πώς να ψαρεύσουν. Η κυρία Γκαμπριάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σιμίτη, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η δημιουργία του καταπιστεύματο για την Αφρική παραμένει καινοτόμα, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά ότι έχουν υπάρξει 11 αναπτυξιακά ταμεία ε, που προηγήθηκαν και δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν ε, την κρίση που ζούμε σήμερα. Θα πρέπει να, λοιπόν να διαρωτώμαστε διαρκώ γιατί. Ε, ναι στη χρηματοδότηση της εφηούς χρηματοδο... Ε, την Εφη, ναι στα αποτελέσματα, καταρχήν ε, ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, αλλά ε, σύνεση θα πρέπει να δείξουμε με multi-buyer, με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτών δωρητών και σκεφτούμε από κοινού πώς αυτό το, το ταμείο θα μπορέσει να έχει παγκόσμια εμβέλεια. Το καταπίστευμα αυτό θα πρέπει να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες αυτών των χωρών πέρα από την επίγουσα κατάσταση, ώστε να προβλέψουμε καλύτερα την επόμενη κρίση. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία λοιπόν αυτών των καταπιστευμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα αναπτυξιακά κονδύλια. Και τέλος τα αποτελέσματα. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, θα πρέπει να πούμε ότι μία από τις δυνατότητες είναι να περιορίσουμε τις προτεραιότητες, ώστε να στοχεύσουμε σε αυτές καλύτερα. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι αμοιβέ υποχρεώσεις των δωρητών και των χωρών εταίρων σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτυχάνονται, χρησιμοποιώντας δείκτες αποδοτικότητας και αναφερόμενες αυτούς διαρκώς αλλά θα πρέπει να, επίσης να δώσουμε περισσότερα για να πάρουμε περισσότερα Έπειτα οι δωρητέ ε, ε, και οι δεσμεύσει του θα πρέπει να ενισχυθούν, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από του Αφρικανού μα εταίρου να κάνουν περισσότερα στη βαλέτα, εάν οι δράσει μα, οι ενεργέ μα δεν αντιστοιχούν στα λόγια μα. Πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπαθίε μα, κομίσοντας τα δέχματα του παρελθόντο. Η μετανάστευση δεν πρέπει να είναι μια θεά ζώνη στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Κυρία Γκαμπριέλ, έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Κόμπορν, τη δέχεστε. Μάλιστα. Κύριε Κόμπορν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ρωτήσω, συμφωνείτε μαζί μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι άχρηστη με τα χρήματα, προφανώς. Έχουμε 20 χρόνια όπου οι υπολογαριασμοί δεν έχουν ε, σωστά ελεγχθεί και δεν έχουν ε, ε, η υπογραφή είναι η χειρότερη υπηρεσία που δίνει βοήθεια στην Αφρική ή όπου στο καλό βρίσκονται αυτοί οι καταβλισμοί στα τουρκικά σύνορα. Δώστε τα χρήματα κατευθείαν οι χώρες και όχι στους καταβλισμούς. Τι, ποιο νόημα υπάρχει να τα δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας βγάλουμε τον, τον μεσάζοντα και θα δώσουμε κατευθείαν στους καταβλισμούς. Συμφωνείτε μαζί μου. Κυρία Γκαμπριέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ερώτησή Σα Δύο στοιχεία έχω να προσθέσω. Καταρχήν πιστεύω ότι αν δεν έχουμε καταλάβει το μέγα δίδαγμα αυτής της κρίσης, είναι ότι ακριβώ θα πρέπει να σκεφτούμε προηγουμένω ότι έχουμε ενεργήσει, αν είχαμε ενεργήσει ω Ένωση εκ των προτέρων, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτέ τι διαστάσεις κρίσης. Στο πρώτο σα ερώτημα, όχι λοιπόν. Και δεύτερον, αρκεί να δούμε τα στοιχεία που δείχνουν πόσο Ορισμένοι δείκτες έχουν βελτιωθεί χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λιγότερη φτώχεια, έχουμε λιγότερα ε, ε, παιδιά που υποσυτίζονται, λιγότερες γυναίκες που είναι χωρίς ε, υγειονομική περίθαλψη. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί σε λίγα χρόνια έχουμε αποτελέσματα. Είτε το θέλετε είτε όχι, η είναι εν τη ενώση. Ο Πρόεδρος, λοιπόν, φαίνεται να διαφωνείτε. Θα τα συζητήσετε αργότερα, διμερώς αν θέλετε. Τώρα το λόγο για ο κύριος Γκερέρο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις προθέσεις και τους στόχους που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των ταμείων. Όλο και πληθαίνουν οι κρίσεις ε, και διαρκούν και περισσότερο. Όλο και πληθαίνουν οι ανάγκες, οι εκτοπισμένοι, αλλά δεν έχουμε μεγαλύτερη και περισσότερη χρηματοδότηση. Ούτε επαρκή για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές. Είναι ε, όλο και πιο απρόοπτη αυτή η χρηματοδότηση, οπότε δεν μπορούμε να φροντίσουμε τον κόσμο που το έχει ανάγκη. Γι' αυτό πιστεύω ότι καλώς να ορίσουν αυτά τα ταμεία αν μπορέσουν να φέρουν περισσότερο συντονισμό, περισσότερη πρόβλεψη, περισσότερη χρηματοδότηση και περισσότερη βοήθεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση. Αλλά μην γελιόμαστε και να μην ξεγελάμε και κανέναν. Περισσότερα χρήματα ε, προέρχονται από άλλα ταμεία, συγκοινωνούν τα δοχεία που είχαν προβλεφθεί για παρόμοιες δράσεις. Και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε, αλλά αν δούμε τον κατάλογο των συνεισφορών των κρατών μελών, δεν θα πω πια ε, κράτη είναι αυτά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν ούτε με τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ούτε με τις ανάγκες του κόσμου. Οπότε, τι θα πρέπει να καταφέρουμε εμείς. Να είναι συμπληρωματικά αυτά τα κονδύλια και όχι υποκατάστατα άλλων ε, προσπαθειών. Αν είμαστε ειλικρινεί, όταν πρεσβεύουμε και κηρύσουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που προσπαθεί να ξεφύγει από την πείνα και τον πόλεμο, θα πρέπει να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη για να γίνουν και τα κηρύγματά μας αυτά όλα πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, η κυρία Επίτροπος θα απαντήσει και σε αυτή την ερώτησή σας. Ε, στο μεταξύ δίνω το λόγο στην κυρία Τρεμπέτσιος. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Προφανώς το πρόγραμμα βοήθειας για τη Συρία είναι ευπρόσδεκτο. Επιτέλους, ε, και ελπίζω ε, να φτάσουν τρόφιμα στους καταβλισμούς. Υπάρχουν πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει τη συνεισφορά στην ύπατη αστεία παρόλο που ε, χτυπούσαν τα καμπανάκια και η γερμανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοούσαν τα προβλήματα. Τώρα προσπαθούν να φέρουν στο πλευρό τους την Τουρκία ε, με μεγάλη γενεοδορία. Η Τουρκία έχει κάνει οπισθοδρόμηση εδώ και τόσα χρόνια στον εκδημοκρατισμό, ελευθεροτυπία, ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντα. Τώρα ο κύριος Γιούνκερ του έταξε και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Τι τον έχει πιάσει τον κύριο Γιούνκερ. Δεν μιλάει με τον Τούσκ Πρόσφατα ο Τούσκ ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και σωστά μίλησε και προειδοποίησε για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Η Ευρώπη θα πρέπει να λύσει τα προβλήματά τη μόνη τη. Είναι παραδοσιακά αυτά καθήκοντα των κρατών μελών, όπω η προστασία των συνόρων. Δεν θα πρέπει να πέσουν θύματα στη χύπικη κουλτούρα Μέρκελ που κυριαρχεί αυτόν τον καιρό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χριστοφόρου, παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κανένας δεν αφισβητεί και δεν διαφωνεί ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη και αλληλεγγύη για το προσφυγικό ζήτημα. Κανένας σε αυτή την αίθουσα πιστεύω δεν αισθάνεται ότι πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη, οι ίδιοι Ευρωπα... Ευρωπαίοι πολίτες είναι οι μοναδικοί που στάθηκαν αλληλέγγυοι για το προσφυγικό ζήτημα. Και το προσφυγικό ζήτημα θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διεθνές ζήτημα. Δεν μπορεί μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδεικνύει ευαισθησία και αλληλεγγύη και όλες οι άλλες χώρες να διαφορούν. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να καταβάλει το άπαντο δυνάμεων της Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξεύρει πόρους να στηρίξει το προσφυγικό και να μην δημιουργείται ένα διεθνές ταμείο στήριξης για το προσφυγικό. Είναι διεθνές θέμα το προσφυγικό που αφορά και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αφορά όλες τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι αραβικέ χώρε να είναι γνωστέ για τα τεράστια επενδυτικά του ταμεία και να μην διαθέτουν ούτε έναν ταμείο, ούτε έναν ευρώ, ούτε έναν πετροδολάριο για να στηρίξουν και αυτή την προσφυγική κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι αδικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πολλοί αναφέρουν ότι δεν έπραξε όσα έπρεπε να πράξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Όμω η μόνη που έπραξε για το προσφυγικό είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ απαράδεκτο και δεν το λέω ούτε από προκατάληψη ούτε για κανένα άλλο λόγο. Θεωρώ απαράδεκτο χώρε όπω η Τουρκία, αντί να πράξει το αυτονόητο για το προσφυγικό όπω πράττουν άλλε χώρε μεσογειακέ και μέχρι και την Ευρώπη είναι ευρωπαϊκέ χώρε, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το προσφυγικό, βάζει μπροστά του πρόσφυγε για να κερδίσει ανταλλάγματα. Για να μην υπενθυμίσω τον ύποπτο ρόλο που διαδραμάτισε και τον καταστροφικό ρόλο για την αστάθεια στην περιοχή και για να δημιουργηθεί το προσφυγικό πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφόρου. Έχετε μια μπλε κάρτα του κυρίου Wolf, συγγνώμη. Τη δέχεστε, κύριε Χριστοφόρου. Yes. Mr. Wolf, you have the floor. I'm great. Κύριε Χριστοφόρου, χαίρομαι που υποστηρίζετε την έννοια ότι δεν είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο. Εγώ έλεγα από καιρό ότι στον ΟΗΕ έπρεπε να τεθεί. Δέχεστε λοιπόν ότι ο, και ο ΟΗΕ έχει παραλείψει πολλά γιατί δεν κάλεσε μια διεθνή διάσκεψη για να συζητηθεί αυτό το θέμα διεθνώς και παρέμεινε μόνος του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Forum, you have the floor. Βεβαίω και συμφωνώ. Δεν είναι μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε δείγματα και πήρε αριστεία όσον αφορά την ελληνική και είμαστε Ένωση Αλληλεγγύη. Γι' αυτό στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό τον λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ναι, ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πρέπει να πάρει πρωτοβουλίε. Και άλλε χώρε οι οποίε σιωπούν αυτή τη στιγμή και δεν είναι το επίκεντρο των συζητήσεων όφυλαν να συνεισφέρουν. Τουλάχιστον οικονομικά δεν μπορούν μεγάλες δυνάμεις από την Αμερικάνικη Ήπειρο, από τις Αραβικές χώρες, από τη Ρωσία και άλλες χώρες να μην συνεισφέρουν και να περιμένουν τα πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό κάνω έκκληση και σαν πρόταση προς την κυρία Αντιπρόεδρο να απευθυνθούμε και σε άλλους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία το προσφυγικό και αν δεν το αντιμετωπίσουν να μείνουν αυτοί εκτεθειμένοι και να μην μένει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτεθειμένη για ένα ζήτημα που έκανε τα πάντα. The next speaker is Mr. Ο έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν ε, ευτυχής που ήμουν νωρίτερα στην Βαλέτα σήμερα. Καλωσόρισα τους Αφρικανούς εκπροσώπους και ευτυχής επίσης που είμαι πίσω εδώ για να καλωσορίσω το καταπίστευμα για τη Συρία. Να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν γι' αυτό και είμαι ευτυχής που το Κοινοβούλιο πρόθεσε το, αυτό το θέμα με την ψηφοφορία στις 18 Οκτωβρίου σήμερα στη διάσκεψη κορυφής και εδώ θέλω να καταστήσω σαφές εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών και των δημοκρατών ότι γνήσια φρέσκα χρήματα θα πρέπει να δοθούν όχι, δεν μπορεί αυτό το καταπίστευμα να στηριχθεί μόνο με την μετακίνηση κάποιων κονδυλίων, εάν θέλουμε θέλουμε να συνοδευτεί και από διεθνείς ε, δωρεές που θα είναι φυσικά εκ οι Βρετανοί συντηρητικοί εκποφελούνται βέβαια αυτή τη συζήτηση για να επικρίνουν την Ευρώπη Διαρκώ Είναι αλήθεια ότι οι αρχικές συμβολές ήρθαν από την Γερμανία και την Ιταλία και όχι από τη χώρα μου, τη Βρετανία. Αλλά πολλοί από εμά στη Βρετανία πιστεύουμε ότι η συντονισμένη βοήθεια μεταξύ των διεθνών δωρητών μπορούν να βελτιώσουν τη βοήθεια για αυτούς που τη λαμβάνουν και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Πρόεδρε, να θυμηθούμε ότι ενώ χιλιάδες πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ευρώπη, υπάρχουν εκατομμύρια στις χώρες γύρω από τη Συρία. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση, αλλά είναι σωστό να σχεδιάζουμε πέρα από την άμεση ανθρωπιστική ανθρωπιστική ανακούφιση και βοήθεια. Πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες αλλά και τις ε, κοινότητες που τους υποδέχονται να τους ε, απορροφήσουν. Η προσφυγική κρίση ε, δεν μπορεί να σταθεί μόνο στην κοντόφθαλμη πολιτική. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ο κύριος Κάρας είναι ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τον κίνδυνο της φυγής μικρότερο από ότι την ελπίδα να επανέλθει η ειρήνη στον τόπο τους. Και ψάχνουν να κρατηθούν από κάπου. Μια ελπίδα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν τους δίνουν ελπίδα και τους τάζουν διάφορα, αλλά λειτουργούν με αμέλεια και επιπολαιότητα. Δύο και δις ε, υπόσχονται και πληρώνουν 100 εκατομμύρια. Αυτά είναι επέσχυντα και επονίδιστα πράγματα. Σταματήστε λοιπόν τα 9,4 δισεκατομμύρια, μην τα δώσετε πίσω. Θα πρέπει να ισοσκελιστούν ε, οι λογαριασμοί, οι προϋπολογισμοί και να γίνουν επενδύσεις για την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση των αιτίων. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε, διότι τα κράτη-μέλη, από ό,τι φαίνεται, τα έχουν χαμένα πλέον. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σπυράκη, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Γεωργίεβα οι έλληνες που υποδέχονται τους πρόσφυγες στη λέσβο και στην Κώ και βλέπουν παιδιά να πνίγονται ταυτόχρονα ρωτάνε τι κάνει η ευρωπαϊκή ένωση για όλο αυτό. η απάντηση είναι ότι η ευρωπαϊκή ένωση κάνει πολλά αλλά συμβαίνει στη ζωή να είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για αυτά που κάνουμε αλλά και για αυτά που δεν κάνουμε και πράγματι εδώ η χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων των ταμείων στην αφρική καθυστερεί δραματικά και το ερώτημα είναι είναι δεσμευτικός ο χρόνος της εθελοντικής συνεισφοράς των κρατών μελών; αρκούν αυτά τα χρήματα; όχι είναι η απάντηση. πότε θα καταβληθούν; κανένας μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει. πώς θα αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση; θα ληφθεί υπόψη ότι δίνονται 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετη πόρη στα κράτη μέλη ώστε να χρηματοδοτηθούν και τέτοιου είδους δράσεις; και τρίτο και πιο σοβαρό πώς παρακολουθούμε ως ευρωπαϊκή ένωση την εφαρμογή των συμφωνιών με τρίτες χώρες οι οποίες χρηματοδοτούνται από δικούς μας πόρους ξεκινώντας από την τουρκία που παίρνει τρία δισεκατομμύρια ευρώ με βάση προταξιακή βοήθεια. πώς το κάνουμε αυτό; πρέπει να δράσουμε. να δράσουμε τώρα. σε διαφορετική περίπτωση ξέρετε ο ευρωσκεπτικισμός θα ανθίζει πάνω στην απελπισία που φέρνουν οι πρόσφυγες στο έδαφος μας. Ευχαριστώ πολύ, η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα σας παρακαλούσα όλους να τηρείτε τους χρόνους σας. Έχουμε καθυστερήσει. Το ξέρω ότι το θέμα μας παθιάζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα τη λύση όσον αφορά την υπέρβαση τη προσφυγική κρίση. Το είδαμε με την υιοθέτηση του σχεδίου προπολογισμού και του διορθωτικού προπολογισμού 7 φέτο. Όμω, οι διορθωτικοί προπολογισμοί δεν είναι ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και τις μη αναμενόμενες εξέλιξεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε πολιτικές προτεραιότητες όταν θα προετοιμάσουμε τον προπολογισμό του επόμενου έτους και να τα σχηματοδοτήσουμε και καταλήλως. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται διαρκώς προετοίμαστη και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις κρίσεις όπως το πάθαμε και το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να καταστήσει σαφέ τα κράτη-μέλη μέσω των διαπραγματεύσεων που κάνουμε τώρα για τον επόμενο προπολογισμό. Πίτροπε Υπουργέ, βασιζόμαστε σε εσά. Θα πρέπει να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στα κράτη-μέλη. Με βάση τα όσα είπε και ο συνάδελφος Κάρας νωρίτερα. Τα δύο αυτά καταπιστεύματα είναι φυσικά σημαντικά, γιατί μόνο βελτιώνοντας την κατάσταση επιτόπου στις χώρες προέλευσης θα καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή την μόνιμη κρίση που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου των ομιλητών, διότι ο κύριος Ριμπέρο δεν είναι εντός της αιθούσης. Περνάμε στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε όλους όσους το ζήτησαν και θα παρακαλώ να σεβαστείτε όμως τον χρόνο σας. Ο κύριος Πόλτσακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν άκουσα το όνομά μου. Γι' αυτό το θέμα θα ήθελα να πω το εξή. Βεβαίω και θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρώπη. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Και δεν θα πρέπει να φοβάται κιόλα η Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να επιδείξει θάρρος. Ε, μιλάμε για δύο ταμεία λοιπόν που ιδρύονται τώρα, δύο καταπιστεύματα για τη Συρία και την Αφρική. Δυστυχώ έχουμε καθυστερήσει όμω. Οι άνθρωποι εδώ και πέντε χρόνια ζουν εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Και αν πιστεύετε ότι ο κόσμος θα κάτσει εκεί να σκοτώνεται ή θα κάτσει σε καταβλισμούς που είναι αναξιοπρεπείς και δεν προσφέρουν κανένα μέλλον σε αυτούς και τα παιδιά τους, δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ ποτέ δεν θα δεχόμουν τέτοιες συνθήκες διαβίωσης και θα ε, έφευγα και εγώ στην προσφυγιά. Πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ η Ευρώπη. Καλωσορίζω αυτά τα δύο καταπιστεύματα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω ότι δυστυχώς έχουν έρθει κατόπιν εορτής. Ο κύριος Φρονζουλίκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εγώ υποστηρίζω το μοναδικό καταπίστευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της Συριακής κρίσης, αλλά και το καταπίστευμα για την αντιμετώπιση των αιτίων ε, της μετανάστευσης και των εκτοπισμένων 5 εκατομμύρια στο 1 και 5,8 εκατομμύρια στο άλλο και ε, θελοντικές δωρεές. Δεδομένο ότι οι αφρικανικές χώρες με ολιγαρχικές ηγεσίες δίγουρα σωστά αυτά τα χρήματα θα πρέπει να μεριμνούμε για τη δαπάνη αυτών των χρημάτων που μπορεί πολύ γρήγορα να εξαφανιστούν λόγω διαφθοράς και ξέρουμε ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αυτές οι χώρες θα πρέπει να τηρήσουν κάποιους όρους και να μην ε, εκβιάζουν κατά κάποιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να πολιτικά να δεσμευθούν για να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση αυτών των καταπιστευμάτων στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το προπολογισμό του 2016. Ευχαριστώ. κύριος Κυρία Τόμασιτ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Τα δύο καταπιστεύματα για τη Συρία και την Αφρική γίνονται από καλή πρόθεση αλλά δυστυχώς δεν θα καταλήξουν σε σωστή διαχείριση του προβλήματος. Είναι μια ακόμη έκφραση ανικανότητας της Ένωσης μπροστά στην κρίση στη Συρία και την Αφρική. Φοβάμαι ότι τέτοια μέτρα στις χώρες αυτές θα είναι αντιπαραγωγικά εφόσον η Ευρώπη δεν ξέρει τι θέλει να κάνει εκεί. Η πρόσκληση που δώσατε στους ε, μετανάστες και πρόσφυγες αντί κατά της θέλησης των λαών μας βέβαια κατέληξε τελικά στο χτίσιμο φραγμών και συμβατοπλεγμάτων μεταξύ γειτόνων. Ποια ακριβώ είναι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Δεν θα έπρεπε πρώτα να το συμφωνήσουμε αυτό και μετά να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε για τους μετανάστας. Πολύ λίγοι από αυτούς προέρχονται από σειράξεις Φοβάμαι ότι πρόκειται για σπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Ο κύριος Γιάκοβιτσιές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος αλλάζει ριζικά μπροστά στα μάτια μας. Και οι διεθνείς σχέσεις επίσης. Και βλέπω τα καταπιστεύματα ως ένα μπάλωμα μεν αλλά που καλό ευπρόσδεκτο είναι και αυτό. Χρειάζεται όμως και άλλη μια νέα πρωτοβουλία που πρέπει να συμπεριλαμβάνει κάτι πιο μακροπρόθεσμο και τους εταίρους μας τους υπόλοιπους και τον ΟΗΕ τους εταίρους μας εκτός Ένωσης που εμπορεύονται μαζί μας και κερδίζουν από αυτό το εμπόριο αλλά δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημα αυτό, ενώ η Ευρώπη έκανε πολλά. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μία, να μία σφαιρικότερη πρωτοβουλία. Γιατί τώρα απλώς βά κάνουμε μπαλώματα για τη Συρία και την Αφρική. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Βίγκας. Ε, ε, θα πρέπει να χωρίς να αγνοούμε τα ανθρωπιστικά προβλήματα, θα πρέπει να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστρέφει καταρχήν και μετά να προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε ε, με ψίχουλα. Είναι συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταστροφή χωρών όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ και, το, και η Συρία. Έχει αίμα στα χέρια της για το θάνατο εκατομμυρίων και για τους πρόσφυγες που εξακολουθούν να φεύγουν από τον πόλεμο και που αντιμετωπίζουν τον κινησμό των θεσμικών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν υπάρχουν αξίες που αιτιολογούν αυτά τα εγκλήματα και η ιστορία θα καταδικάσει τους ηγέτε αυτών των χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπουν να δολοφονείται τόσο κόσμο. Ο κύριος Τάραντ είναι ο τελευταίο ομιλητή, Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν η μετανάστευση είναι πρόβλημα, ίσως θα πρέπει να δούμε την ιστορία ο Homo sapiens από στην, ε, ξεκίνησε από την Κένια και μετά ε, κατέκτησε ολόκληρο τον πλανήτη μας. <laughs> Δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Η κυρία Γεωργίευα πιστεύω κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την κατάσταση. Όμως... Όμως ποτέ δεν θα λυθεί το πρόβλημα απλά δίνοντας περισσότερα χρήματα εκεί στη, στα μέρη όπου βράζει η κατάσταση. Πρέπει να θυμηθούμε την, ε, να σκεφτούμε την ασφάλεια, να σκεφτούμε και να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι χρειαζόμαστε κοινή ασφάλεια άμυνα και εξωτερική πολιτική. Ευχαριστούμε κύριε Τάραντ. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται το κατσδιά και σας ευχαριστώ για την πειθαρχία σα που συμβαστήκατε δηλαδή το χρόνο αγόρευσή σα Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο. Παρακαλώ κυρία Γεωργίβα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσει έχω να κάνω. Η μία είναι ότι πρόκειται για παγκόσμια κρίση και ότι όντως απαιτείται ε, παγκόσμια απάντηση. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε το 20% της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά 50% και παραπάνω ε, σε σχέση με την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Κάνουμε δηλαδή αυτό που μας αναλογεί και είναι σημαντικό και όσοι μπορούν να συμβάλλουν θα πρέπει να το πράξουν. Περισσότερη ε, σπλούτο σημαίνει περισσότερες ευθύνες. Πρέπει να καλέσουμε σε κινητοποίηση ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να βοηθηθεί. Με τον ίδιο τρόπο που η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μας έδειξε ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά για να οικοδομήσουμε θεσμούς και δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά αυτή την κρίση, το ίδιο και η προσφυγική κρίση που εκθέτει κάποιες από τις ελλείψεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όσον αφορά τη συλλογική δράση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα δούμε προτάσεις από... Μάλλον για... Ε, ε, συνοριακούς ελέγχους για την ε, άμυνα και την ασφάλεια στα σύνορα, αλλά πιο σημαντικό είναι πιο συντονισμένη και συνεπτική ε, μέσο και μακροπρόθεσμη συνεργασία με τις χώρες που χρειάζονται τη βοήθειά μας για να μπορέσουν να οικοδομήσουν τις δικές τους δυνατότητες και να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές τους προκλήσεις. Και βέβαια εννοείται ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση είναι καταρχήν να μην υπήρχε. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην πρόληψη των σειράξεων, στην επίλυση των ε, συγκρούσεων, ώστε να ε, λιγότεροι άνθρωποι να επηρεάζονται στο μέλλον από αυτό που θα ε, από όλα αυτά γιατί και οι κλιματικές αλλαγές θα φέρουν και άλλες μετακινήσεις και φυσικά οι βίες σειράξεις οδηγούν τον κόσμο στην προσφυγιά. Και ναι, δεν είμαστε τέλειοι, αλλά ναι, είμαστε ακόμα πιο δεσμευμένοι και συμβάλλουμε πολύ περισσότερο από ότι πολλοί άλλοι γύρω μας. Και έπειτα κάποιες πιο συγκεκριμένα σχόλια. Τονίστηκε ότι πρέπει να στραφούμε προς άλλους ε, εταίρους κλειδιά στην ανάπτυξη και βοήθεια. Και το κάνουμε. Εγώ την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στη ΗΠΑ για να συνδεθώ με την Παγκόσμια Τράπεζα του Δουνουτού και την Αμερικανική κυβέρνηση που είναι ο πιο σημαντικός μας εταίρος για το πώς θα προσεγγίσουμε αυτές τις κρίσεις και χρειάζεται να επεκταθούμε πέρα από την άμεση επίγουσα ανταπόκριση για να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες ώστε οι χώρες να έχουν έναν περιθώριο απέναντι στις κρίσεις ώστε η, η παγκόσμια κοινότητα να ευθυγραμμιστεί στο πώς αντιμετωπίζουμε την ευαισθησία αυτή. και με χαρά βλέπω ότι το δούνο του φτιάχνει πολύ πιο ισχυρές δαμές ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ευάλωτες χώρες. Και είναι λάθος μου που δεν ξεκίνησα λέγοντας ότι τα 2,3 δις θα τοποθετούμε σε ένα πλαίσιο αυτού που είναι τώρα 10 δις από την Κομισιόν για να αντιμετωπιστεί η προσωπική κρίση εντό και εκτός. Η ιδιαιτερότητα αυτών των καταπιστευμάτων είναι ότι είναι ένας νέος τρόπος για να οργανώσουμε καλύτερα και να αναπτύξουμε καλύτερα τους σπόρους μας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά αυτό δεν μειώνει τη ε, ε, λογοδοσία. Ε, και φυσικά θα σας πούμε τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ελπίζω πως θα είναι και πιο ουσιαστική η συνεργασία γιατί θα είναι με, βάση ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα γιατί απλά ανακατατάσσουμε τόσα ήδη υπάρχουν στον προπολογισμό μας. Το η απάντηση είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα είναι φρέσκα χρήματα. Έχουμε πάρει ένα δις από το αποθεματικό του Αναπτυξιακού Ταμείου. Είναι χρήματα δηλαδή που τώρα προστίθενται για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κρίση. Και επίσης έχουμε κάνει κάποια ανακατανομή χρημάτων από δραστηριότητες μικρότερης προτεραιότητας. Ε, και νομίζω πως αυτό σωστά το πράξαμε. Επικριθήκαμε και δυστυχώς αυτοί που επικρίνουν ήταν εδώ για να τα πούνε, αλλά τώρα δεν ακούν την απάντηση. Κανονικά όταν θέλεις μια ερώτηση πρέπει να περιμένεις και την απάντηση. Εν περιπτώσει, εμείς έχουμε ένα πολύ καλό ρεκόρ ε, όσον αφορά τα αναπτυξιακά μας προγράμματα και ιδιαίτερα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μας έχει τοποθετήσει ως τους πρώτους σε αυτή την ε, περίπτωση και είμαι πολύ περήφανη γιατί εκεί ήμουν προηγουμένως και γι' αυτό γιατί είμαστε χρόνια επιτόπου και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι προτεραιότητες. Έχουμε αναπτύξει δε τους πόρους μας σε 8 ανθρώπους ανθρώπους στη Συρία ε, αυτό όμω δεν είναι σωστό. Ε, δεν... Μας είπαν ότι δίνουμε όλα τα χρήματα στι γειτονικέ χώρε, αλλά όχι. Δεν είναι αλήθεια. Τα μισά πάνε στη Συρία και μάλιστα σε περιοχέ που κρατώνται στις, ε, από του ε, επαναστάτε, που ελέγχονται από του επαναστάτε. Είμαστε από του λίγου που ποτέ δεν εγκαταλείψαμε αυτού που πλήττονται περισσότερο στη Συρία, εκεί που δηλαδή πέφτουν βόμβες και όπου ο κόσμος βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Επίσης υπόθηκε αρκετές φορές ότι σπαταλούμε τα χρήματα και ότι οι λογαριασμοί μας δεν έχουν ε, ε, πάρει απαλλαγή εδώ και 20 χρόνια. Όχι, λάθος. 8 χρόνια τώρα έχουμε πάρει την απαλλαγή και μάλιστα εχθές μόλις πήραμε την τελευταία απαλλαγή. Δεν πρέπει λοιπόν να μπερδεύουμε σφάλματα τα οποία είναι ανεπιθύμητα αλλά προς, ε, γι' αυτό πρόκειται, δεν πρόκειται για ε, σπατάλη, ούτε για απάτη. Ε, πολλές φορές σφάλματα μπορεί να συμβούν και πρέπει να είναι επίσης σαφές ότι ναι, αντιμετωπίζουμε μια τεράστια, τεράστια πρόκληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά αν συνεργαστούμε. Έχουμε σχεδιάσει μια νέα πλατφόρμα για δράση όπου θα έχουμε περισσότερες συμβολές από τα κράτη-μέλη αλλά και από άλλους. Και υπήρξαν κάποια θερντικά σημάδια από τη ΣΥΠΑ ας πούμε ότι μπορεί να μπουν και εκείνοι στο καταπίστευμα για τη Σύρια είτε άμεσα είτε παράλληλα θα δούμε. Ε, πάντως θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Κοινοβούλιο που ασχολείται με αυτό το θέμα για την έκκληση που κάνετε για περισσότερα κοινή δράση από πλευρά των κρατών ε, ε, και θα κλείσω ευχαριστώντας σε όλους ιδιαίτερα στο Λουξεμβούργο τον Υπουργό Σμιτ Μακάρι όλοι να δούλευαν σαν και εσάς. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γεωργίευα, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την απάντηση. Δίνω το λόγο στον Υπουργό. Κύριε Σμιτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω εγώ. Στο είπε μόλις η, κυρία Αντιπρόεδρος. Η κατάσταση επήγει απολύτως και τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιήσουμε τους πόρους που μας χρειάζονται. Εντάξει, γεγονό γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί ακόμα να μην έχουν αντιδράσει παρκώς. Μπορεί να μην έχουν ανταποκριθεί σε όλες τους τις υποσχέσεις. Ακόμα. Πάντως σήμερα εκπέμψατε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο εγώ φυσικά θα διαβιβάσω έτσι ώστε τα κράτη να σεβαστούν και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά να πούμε ειλικρινώς ότι δεν είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι δύο ενότητες, οι οντότητες. Από τη μια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με το προϋπολογισμό της και από την άλλη τα κράτη-μέλη με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τους κρατικούς. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μπορεί κάποια χρήματα να προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά είναι και των κρατών μελών και άλλα χρήματα να έρχονται από άλλες πηγές. Κοινό είναι ο Κουρβανάς, σε περιπτώσει. Και τώρα μιλήσατε και για το καταπίστευμα. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε δίκιο και οι υπόλοιποι και οι βουλευτές που το είπαν. Το θέμα αυτό αφορά κατά πρώτο λόγο την Ευρώπη, διότι όλα αυτά συμβαίνουν στην άμεση γειτονιά μας και μας αφορά, γιατί στην Ευρώπη έρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ευρώπη. Η κρίση αυτή είναι διεθνής. Άρα, είναι προφανέστατο ότι εάν θέλουμε να δράσουμε, θα πρέπει ε, να ε, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια σύνολη η διεθνής κοινότητα και μάλιστα χώρες που έχουν κάθε συμφέρον να αντιμετωπιστεί σωστά η κρίση. Δεύτερο, ε, το πιο μακροπρόθεσμο βεβαίως έχει να κάνει με την ανάπτυξη, έχει να κάνει και το πώς θα σχεδιάσουμε ξανά τις αναπτυξιακές μας πολιτικές, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τρομερή επιτυχία όλη αυτή η πολιτική, ούτε απόλυτη να δούμε πού ε, πηγαίνουν τα χρήματα, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στις δαπάνες αυτές, πώς μπορούμε να φέρουμε ενώπιον των ευθυνών τους αυτές τις χώρες, αν μπορούμε, γιατί είπατε μερικοί από εσά ότι ε, πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε καν κρατική υπόσταση, για να μην μιλήσω για κράτος δικαίου. Ας πούμε, μιλάμε για την Ερυθρέα. Και υπάρχει ένα καθεστώς που οδηγεί τους νέους ε, στο να τραπούν στη φυγή. Γιατί ε, αλλιώς θα περάσουν όλη τη ζωή ε, σε ένα στρατό τον οποίο απορρίπτουν. Είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση λοιπόν και χρειάζεται και πιο μακροπρόθεσμη δράση. Συμπέρασμα από τη συζήτηση αυτή που ήταν τόσο πλούσια ότι θα πρέπει να στείλουμε σαφές μήνυμα η μόνη λύση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα είναι μια λύση αλληλεγγύης. Αυτή και καμία άλλη. Ούτε να ποντάρουμε στον έναν ή στον άλλον, ούτε να κάνουμε απόσυμασματικές και κατακαιρματισμένες δράσεις. Δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Αυτό εγώ κρατώ από τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.